Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση μας. Ε, καθυστέρησα επειδή είχα συνάντηση με ε, οργανώσεις γεωργών από την Τσεχία και Σλοβακία. Από τις 8 ήμουν ε, σε συνάντηση με τέτοιες οργανώσεις και άκουσα και την παρέμβαση του Τσέχου Υπουργού Γεωργίας ε, να με συμπαθάτε για αυτή την καθυστέρηση, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσουμε ε, το χαμένο έδαφος. Ας πάμε στην ημερήσια διάταξη λοιπόν. Όπως ξέρετε, Ε, είχαμε δύο ψηφοφορίες. Ε, μία κατέπεσε, αλλά την άλλη την ψηφοφορία θα την κάνουμε για τα εγωπρόβατα. Δεν έχει... Ναι, ναι, για τις πρωτεΐνες δεν θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε μόνο για τα εγωπρόβατα. Όπως ξέρετε, απεβίωσε ο συνάδελφος, ο κύριος Εντουάρ Φεράν. Πρόωρα χάθηκε ο συνάδελφος. Ε, εργαζόταν εδώ και συνεργαζόμασταν ε, για πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν πολύ προσιλωμένος και αφοσιωμένος ε, στη γεωργία, στους γεωργούς και πολύ δραστήριο μέλο, μέλος της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ε, στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας ε, στους, στους συγγενείς, οικείους φίλους τους, στις πολιτικές ομάδες. Ήταν πάντα ανοιχτός, συνεργάσιμος, χαμογελαστός, μπορεί να μην συνέπταν πάντα οι απόψεις μας. Αλλά με τέτοια ανταλλαγή απόψεων προσπαθούσαμε όλοι να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον των Γεωργών και της Γεωργίας. Ο καθένας με τις δικές του απόψεις και τις δικές του εκτιμήσεις ε, προσπαθούσε να υπερασπίσει τα συμφέροντα των Γεωργών. Παρακαλώ λοιπόν να σηκωθούμε και να τηρήσουμε ενός λεπτούς υγιής μνήμην εδώ Φερόν. Ευχαριστώ. Ε, μην ξεχνάτε ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας είπα ότι από τις ψηφοφορίες που είχαμε η μία έχει αναβληθεί. Η ψηφοφορία για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες αναβάλλεται. Οπότε περνάμε κατευθείαν στο σημείο 4 που είναι η εκλογή του τέταρτου αντιπρόεδρου της Επιτροπής ε, αφού έμεινε καινή η θέση του κυρίου, ε, ε της κυρίας ε, θα ήθελα να μεταβιβάσει ο συντονιστής και ε, τα συγχαρητήρια της ομάδας και την, ε, τις ευχές για καλή επιτυχία α, ε, της κυρίας Δαντσίλα στο νέο έργο της. Είναι για μας μεγάλη τιμή για την Επιτροπή Γεωργίας που πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας έγινε πρωθυπουργό της χώρας της κυρία Δαντσίλα. Της είχαμε εκφράσει και τις προσωπικές μας ευχές και τα συγχαρητήρια. Όπως είπε λοιπόν περνάμε στο σημείο 4 γιατί θα πρέπει να εκλέξουμε επίσημα τον τέταρτο αντιπρόεδρο, μια και έμεινε κενή η θέση του αντιπρόεδρου μετά την αποχώρηση της κυρίας Νταντζίλα. Οι πολιτικές ομάδες ε, μπορούσαν να υποβάλουν τους υποψηφίους τους ή και με μονομένοι βουλευτές εφόσον συγκέντρωναν τον απαραίτητο αριθμό. Ο, κύριος την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή υποψηφιότητων. Ο κύριος Αντρίε που είναι ο συντονιστή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα μας κάνει την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα ε, λόγια σας που είπατε. Ντεζίλα, θα ήθελα να πω, σας συντονιστή των Δημοκρατών, ότι χρειάζεται και αντανζήλε πολλά, πολύ, πολύ θάρρος για τα νέα καθήκοντα που ανέλαβε σε μια στιγμή που είναι κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ούριο άνεμο της εύχομαι. Ήταν ενεργό μέλος της πολιτικής μας ομάδας που προωθούσε την Ευρωπαϊκή Γεωργία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας με πεποίθηση και με δύναμη. Θα ήθελα όταν ψηφίσουμε νέο αντιπρόεδρο εν ονόματι των Σοσιαλδημοκρατών την Καμπρίλα Ζωάννα να παρουσιάσω που διαδέχεται τη συνάδελφο είναι πίσω μου για να καλύψει τη θέση αντιπροεδρού της Επιτροπής Γεωργίας με την πεποίθηση ότι τα μέλη αυτής της Επιτροπής θα δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτό το νέο μέλος του Κοινοβουλίου που έχει όλα τα πετούμενα προσόντα τόσο ώστε να εκτελέσει την αποστολή μέλους του τομέα της Γεωργίας αλλά και τα καθήκοντα του Προέδρου. Ευχαριστώ και Πρόεδρε ε, που λαμβάνετε υπόψη αυτή την υποψηφιότητα της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έκερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του τον κύριο Μάρκο Ζούλο, προτείνω. Ο κύριος Μάρκο Ζούλο ε, ήταν συνεργάτης επίσης και πλήρες μέλος της Επιτροπής. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του και οι δύο υποψήφοι είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο για να υποβάλει άλλη υποψηφιότητα, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Νίκολσον ζήτησε το λόγο. Η κυρία Εράς. Όταν ξεκινήσαμε ε, με την ε, συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, είχα ένα πρόβλημα με την διερμηνία. Κατάλαβα ότι ε, δεν θα ψηφίζαμε. Αλλά θα ήθελα να συζητήσω αύριο, στην αυριανή ημερήσια διάταξη, να κάνουμε μια αλλαγή. Και το σημείο 13 να συζητηθεί στη θέση του 12 και το 12 στη θέση του 13. Να γίνει μια αντιστροφή της σειράς δηλαδή μεταξύ των σημείων 12 και 13. Το συζήτησα με τη γραμματεία και μου είπε ότι αν κανένα άλλος δεν έχει αντίρρηση, δεν υπάρχει πρόβλημα με την αλλαγή. Δηλαδή το σημείο 12 ε, να συζητηθεί μετά το 13. Και το 13 του κυρίου Ντόρφμα δηλαδή να συζητηθεί στη θέση του 12. Μια αντιστροφή των δύο σημείων δηλαδή. Ε, Μάλιστα. Οι εισηγητέ, δηλαδή ο συντάκτη γνωμοδότη ο κύριος Κάρθη και ο εισηγητή ο κύριος Ντόφμαν συμφωνούν με την αλλαγή, την αντιστροφή αυτών των σημείων το 12 και 13 τη ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Γκάρθη που έχει το 12 συμφωνεί, οπότε θα ακολουθήσει τη συζήτηση του 13, το 12. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω, να κάνω, να ρωτήσω κάτι ενημερωτικό και να ξεκινήσω ε, από την αρχή της Επιτροπής ε, και το πώς συστάθηκε με το σύστημα αντεχών, το EFTD δεν ε, είχε δικαίωμα στην Προεδρία εδώ στην Επιτροπή. Δυστυχώ δεν πέρασε αυτή. Και τώρα πώ βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το σύστημα DONT. Θα ήθελα ένα μέλο της Επιτροπής ε, να είναι βάση του συστήματος DONT και αυτό θα θέλω να το τονίσω γιατί μπορεί να γυρνάω, αλλά αν δεν με πατάει η μνήμη μου, η μνήμη μου θυμάμαι ότι τότε είχε γίνει ένας καυγάς σε ό,τι αφορά το εκπρόσωπο του EFTD που δεν είχε υποστηριχθεί από την Επιτροπή και έτσι οι σοσιαλιστές πήραν την επόμενη αντιπροεδρία. Θα ήθελα μόνο να το διευκρινίσω. Ποιες είναι στην παρούσα φάση οι προδιαγραφέ βάσει του συστήματο DONT. Αυτό, απλά θα το ερώτημα. Proszę o wyjaśnienie pana Παρακαλώ, ο γραμματέα θα το μα εξηγήσει. Κοιτάξτε, το θέμα είναι δύσκολο. Το μόνο που έχω να πω, το μόνο που έχω να πω είναι το εξή. Έχουν γίνει διευθετήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, είτε βάσει συστήματο DONT, είτε όχι. Αυτό είναι αποκλειστικά στο, στην αρμοδιότητα των πολιτικών ομάδων από πλευρά κανονισμού, σε τελική ανάλυση, αυτό που έχει σημασία είναι το τι γίνεται την ημέρα τη εκλογή. Τώρα λοιπόν γίνεται μια ψηφορία, μια εκλογή αντιπροέδρου. Δεν μπορώ να προκαταβάλω το αποτέλεσμα της εκλογής και αυτό είναι που μετράει. Θα πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρέ διαδικασίες και φυσικά δεν μπορώ να σχολιάσω το αποτέλεσμα ενδεχομένω. Ούτε μπορώ να σχολιάσω τι πολιτικές συμφωνίες ενδεχομένως έχουν γίνει εκ των προτέρων. Λυπάμαι. Ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ εθετήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, θα ήθελα απλά να αναφέρω το εξή. Στην ε, ομάδα του Άλντε των Φιλελευθέρων δεν θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοια πολιτική συμφωνία πλέον. Δεν υφίσταται. Και αυτό ήταν σαφέ όταν ε, εκλέξαμε τον Αντιπρόεδρο της Ολομέλειας ε, του Κοινοβουλίου, στη Σύνοδο της Ολομέλειας, ο Αντιπρόεδρος ε, υποτίθεται ότι θα ε, ήταν η Γκεσίνερ Μάισνερ από τις φιλελεύθερους, αλλά η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ψήφισε και μάλιστα μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε υπέρ του υποψηφίου του EFTD. Άρα δεν υπάρχει πολιτική συμφωνία και εμείς είχαμε το τέτοιο ερωτηματικό όπως ο κύριος Νίκολσον και γι' αυτό θα απόσχουμε. Όχι επειδή είμαστε αντίθετοι με τον υποψήφιο, αλλά δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πλέον πολιτική συμφωνία και άρα δεν ξέρουμε αν ε, καλά θα κάναμε να ακολουθήσουμε το σύστημα DONT ή κατά πόσον υφίσταται υποψία πολιτικής διευθετής και συμφωνίας. Αυτό ενημερωτικά για να σας εξηγήσω γιατί θα απόσχουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Να προτείνω το εξή. Οι σοσιαλιστές να κοιτάξουν τι σημαίνει η λέξη σοσιαλιστές Ίσο και δίκαιο μερίδιο. Ίσο και δίκαιο μερίδιο, λοιπόν. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, λοιπόν, θα το δώσουμε σε μία μικρή ομάδα, γιατί δεν υπάρχει ίση και δίκαιη κατανομή στην παρούσα φάση. Μάλιστα, χρήσιμη ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Αλλά και η μέθοδος εντεόντ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην ε, ψηφοφορία. Γι' αυτό περάσουμε στην ψηφοφορία. Να ελέγξουμε καταρχήν ε, τα μέλη της κάθε πολιτικής ομάδας ε, ή να τσεκάρουμε αν κάποιος αναπληρώνεται εδώ στην ψηφοφορία. Κύριε Ντελέα, αντικαθιστά τον κύριο Μέλο. Ο κύριος Μπογκόβιτς την κυρία Πετήρ και ούτω καθεξής. Έχουν δηλώσει οι πολιτικές ομάδες ε, ποιοι αντικαθίστανται για την ψηφοφορία. Γιατί μερικές φορές ε, κάποιοι αναπληρωτές θα ψηφίσουν στη θέση των τακτικών μελών που απουσιάζουν. Αλλά τα έχουν κανονίσει οι ομάδες. Έχουμε δύο υποψήφοι που δέχτηκαν ε, τις Έχουμε δύο υποψηφίους που συμφώνησαν με την υποψηφιότητά τους τους κυρίους Ζωνάν και Ζούλο. Τσούλο. Ε, μάλλον την κυρία Γκαμπριέλ ε, Ζέναν και τον κύριο Τσούλο. Με το πράσινο κουμπί ψηφίζετε την πρώτη υποψήφια, με το κόκκινο τον δεύτερο, τον κύριο Τσούλο. Ε, όποιος δεν συμφωνεί με κανέναν μπορεί να κρατήσει αποχή. Να επισημάνω ότι υπάρχει ένα θέμα ε, με την διερμηνία, ένα τεχνικό ζήτημα. Και η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Είναι σημαντικό. Κάθε λέξη να μεταφέρεται σωστά. Ιδάλω θα χαθούν κάποια στοιχεία και λυπάμαι. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να πω από πλευρά τη ομάδα μα ότι συμφωνούμε με τον υποψηφίο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επαναλαμβάνω. Όσοι ψηφί, θέλουν να ψηφίσουν την κυρία Ζωνανό, θα πρέπει να πατήσουν το πράσινο κουμπί. Όσοι ψηφίζουν τον κύριο Τσούλο, πατούν το κόκκινο κουμπί. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Και παρακαλώ, οι συντονιστές των ομάδων να ελέγξουν ε, τον αριθμό των ευρωβουλευτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αν ε, αποσιάζουν κάποια τακτικά μέλη, ποιοι αναπληρωτές τα αντικαθιστούν στην ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία, επαναλαμβάνω. Πράσινο κουμπί για την υποψήφιο των σοσιαλιστών, κόκκινο για τον κύριο Τσούλο. Άρχεται ψηφοφορία. Oh, μου Συγγνώμη, πρέπει να βάλουμε και την κάρτα βέβαια. czy jeszcze w tej chwili można dokonać Μπορείτε μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνετε αλλαγέ στο μέτρο που δεν έχω κηρύξει το πέρα τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έχουμε μία ψήφο του σοσιαλιστών παραπάνω. Okay, now. It is not Καλώς, εντάξει. Όλα εντάξει τώρα, έτσι. Ωραία. Δεν έχουμε υπεράριθμους. Οπότε κλείνει, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ετοιμάστε τα αποτελέσματα. Συγχαίρουμε την κυρία Γκαμπριέλα, την υποψήφια των σοσιαλιστών, που ε, θα είναι η τέταρτη αντιπρόεδρος Επιτροπής και την καλούμε να αναλάβει τη θέση της. Υπάρχει θέση δίπλα στο γραμματέα μας, τον Φιλίπ. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Συγχαρητήρια και πάλι στη νέα μας αντιπρόεδρο αμέσως θα δώσω το λόγο στην κυρία Ράς Γκαρσία πριν ψηφίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της για την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και πάρα πολλές τροπολογίες, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η εισηγήτριά μας, η κυρία Εράς Γκαρσία. Παρακαλώ, κυρία Γκαρσία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η έκθεση αυτή αφορά ένα πολύ ευαίσθητο τομέα, το τομέα εγωπροβάτων. Είναι ένας κλάδος που τις τελευταίες δεκαετίες σημείωσε πολύ μεγάλες ε, ζημίες και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στην Επιτροπή ότι αξίζει αυτή την ιδιαίτερη προσοχή που το αφιερώνουμε. Κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες για μια έκθεση που είναι έκθεση πρωτοβουλίας που κανονικά δεν ε, συγκεντρώνει ε, τόσε τροπολογίε. Και αυτό δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον τη Επιτροπή μα για το κλάδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τι πολιτικέ ομάδε, ε, του συνεργάτε, το προσωπικό, τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πραγματικά είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία. Και ε, καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε αρκετές συμβαστικές τροπολογίες και για το διατακτικό και για τις αιτιολογικές σκέψεις. Και θεωρώ ότι ε, η ψηφοφορία θα είναι πολύ πιο ομαλή από ό,τι αναμέναμε. 18 συμβαστικές τροπολογίες έχουμε συντάξει για το νομοθετικό κείμενο και 7 πλέον συμβαστικές τροπολογίες για τις αιτιολογικές σκέψεις. Αυτά δείχνουν ε, τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να διεξαχθεί πιο ομαλά και γρήγορα η ψηφοφορία και να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη γνώμη. Ελπίζω να μην υπάρχουν προβλήματα με την ψηφοφορία και τον κατάλογο ψηφοφορίας. Είχαμε μέχρι τελευταία στιγμή κάποια μικρά προβλήματα. Λυπάμαι που τελευταία στιγμή μόνο οριστικοποιήθηκε ο κατάλογο ψηφοφορία και το μοιράσαμε, αλλά ακριβώ επειδή είχαμε προβλήματα μέχρι τελευταία στιγμή καθυστερήσαμε κάπω. Και μάλιστα μερικέ ε, τροπολογίε μπορούμε να τι ψηφίσουμε ομαδών. Για παράδειγμα, τι συμβαστικέ τροπολογίε 15, 16 και 17, γιατί συμφωνούμε όλοι ω προ αυτό αυτά. Ελπίζω να πάει καλά η ψηφοφορία και στην ε, Ολομέλεια να υπερψηφιστεί η έκθεση, γιατί παραλαμβάνω αξίζει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίζει αυτό ο κλάδο. Και μάλιστα θα πρέπει να τον προσέξουμε εν ώψη των μελλοντικών μα εμποριών συμφωνιών που μπορούν να τον θέσουν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία και αν χρειαστούμε και άλλη βοήθεια, θα σα ρωτήσουμε, κυρία Γκαρσία. Ψηφίζουμε τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με δύο ψήφους διαφορά μόνο. Οπότε είχε νόημα που κάναμε τον έλεγχο. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία... Α, συγγνώμη. 284. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 145. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146. 146. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καλώ το ελέγξαμε. 322. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 365. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 153. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 160. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 ή μάλλον πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 381 Το κύριο Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 72. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 173. Και η 323 που είναι πανομοιότυπη υπέρ. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 177. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με την ίδια διαφορά. Αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. 177. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. 178. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Εγκρίνεται. 190, μάλλον όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 4, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 195 του κυρίου Νταντάν. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 196. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Εγκρίνεται. 204 και 200, ή μάλλον όχι, 204 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 207 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται τροπολογία. 216 δεκαέξι. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 356. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 194. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 194 άρχεται η ψυχοφορία Yes, 194. Zamykam, zamykam. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 219 λέει ο πρόεδρος, υπέρ κατά απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά απορρίπτεται. 386 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 229. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 203 υπέρ. 230 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 238. Ή μάλλον πρώτα, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 236. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 238 υπέρ κατά δεν σηκώνατε εμφανώς τα χέρια σας ε, για την 238 οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά Τροπολογία 370. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 385. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 248 υπέρ. Εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν ξέρω τι ψήφισε ο κύριος Αντρία. 2.52, άρχεται ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Αλλά δεν ήταν σαφές. 253. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 253 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται οριακά με μία ψήφο διαφορά. 256. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία ή μάλλον 274. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 264. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 265 υπέρ εγκρίνεται. 267. 267. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 285. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 294. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 380 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 383. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 383 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Άρχεται ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 12. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 305. Νόιχλ και Ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 306. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Εγκρίνεται. 309 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 321 της κυρίας Νόιχλη, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και περνάμε στις συμβαστικές 15, 16 και 17, από κοινού τις ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τρεις συμβαστικές τροπολογίες 15, 16 και 17. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Και πάμε στην 371. Σε κύριο Τσούλο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 320. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 325. Ποιος είναι υπέρ. Η 320 εγκρίθηκε. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 320. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 325. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 249. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 249. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Μπράβο σας. Καλά που το ελέγξαμε. 251 εγκρίνεται. 215 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 382 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και πάμε στην 330 τροπολογία της κυρία Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 375 υπέρ. Εγκρίνεται. 376 υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε καλοκακού. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 376. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μπράβο σας. 219. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Εγκρίνεται. 372 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 373 υπέρ εγκρίνεται. 254 υπέρ κατά απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κυρία Νόιχλ και κύριε Ταραμπέλα. Εγκρίθηκε η τροπολογία σας. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 1. Α, ή μάλλον, α, άρχεται η α Ένα λατινικό συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 14 του κυρίου Νέκοφ. Υπέρ εγκρίνεται. 16 υπέρ εγκρίνεται. 17 υπέρ εγκρίνεται. 18 ποιος είναι υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 23, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. μπράβο σας. Συμβαστική τροπολογία 2, λατινικό, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 25. Όχι. 26. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 27, η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3, λατινικό, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 39. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Εγκρίνεται. 56 υπέρ εγκρίνεται. 57 υπέρ, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 61. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 63. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Εγκρίνεται. Με την ίδια διαφορά. 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 67. Άρχεται η ψηφοφορία. για την 67. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Εγκρίνεται. 73 υπέρ εγκρίνεται. 74 υπέρ εγκρίνεται. 75 υπέρ εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά απορρίπτεται. 78 υπέρ εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 92. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 95 υπέρ, εγκρίνεται. 96 υπέρ, εγκρίνεται. 98 υπέρ, εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 101 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Μπράβο σας. 105. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 λατινικό. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110. Τέλος ψηφοφορίας και όντως εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω ότι ψήφισε ο κύριος Αντρία. Ας το ελέγξουμε λοιπόν καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 111. Γιατί πρώτα κοιτάω τους συντονιστές Τη ε, οδηγία δίνουν και μετά κοιτάω την ομίγυρη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 112 ήταν αυτή. 113 και 114, 115 και 116 είναι παρόμοιες, ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο και για αυτές. Καλώ σας το ελέγξουμε παρόλο που θεωρώ ότι εγκρίνονται. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Περιμένουμε να αλλάξει την κάρτα του ο κύριος Γιάρ. Είστε έτοιμος, κύριε Γιάρ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117 άρχιτη ψηφοφορία. 117. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 122. Του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 124 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 125. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση του σχεδίου ψηφίσματος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψηφίσμα. Συγχαρητήρια κυρία Ρας Γκαρσία, έχετε το λόγο. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξή σας Ευχαριστώ εκ μέρου του κλάδου. Είναι πολύ σημαντικό. και αυτό και ελπίζω και στο, στην Ολομέλεια να έχουμε ε, τέτοια πλειοψηφία ώστε να υπερψηφίσουμε το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση, γιατί πραγματικά αξίζει να ανθίσει ο τομέα των εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε και πάλι κυρία Γκαρσία και ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Ε, Φίλιπ break Ο Φιλίπ θέλει μια δίλεπτη διακοπή, ένα δίλεπτο διάλειμμα. Το επόμενο μα θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό, το πρασίνισμα που λέμε, το greening. Και ίσω θα περιμένουμε αλλαγή στο θέμα αυτό στην επόμενη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ μετά το 2020. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Σάμο Γέρεπ, μέλος του πρώτου τμήματος ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα μας παρουσιάσει την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τον οικολογικό προσανατολισμό και την πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής ε, αυτού του νέου συστήματος. Έχαμε πολλές προσδοκίες από τον οικολογικό προσανατολισμό και έχουμε και τη νέα οικολογική ενίσχυση, που είναι ένα νέο είδος άμεσης ενίσχυσης ε, που θεσπίστηκε το 2013 με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Οι πρώτες ενισχύσεις ε, δόθηκαν το 2016. Ε, το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις επιζήμιες επιπτώσεις στις γεωργικές πρακτικές, ιδιαίτερα της εντατικής γεωργίας και πώς επηρεάζουν το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Σάμο Γέρεπ στα πλαίσια αυτής της ειδική έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, με ενδιαφέρει και εμένα ιδιαίτερο σε αυτό το θέμα του οικολογικού προσανατολισμού γιατί είναι ιδιαίτερα επίμαχο και αμφιλεγόμενο. Ήδη περιμένω πώς και πώς ε, την παρέμβαση του κυρίου Ντες για τον οικολογικό προσανατολισμό. Ο κύριος Δες και ο κύριος Δεκάστρο κατάφεραν να περάσουν κάποιες τροπολογίες για το θέμα αυτό στον κανονισμό Omnibus. Θα μας τα πω αργότερα. Πάντως, ε, η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου θα μας βοηθήσει στις ε, μελλοντικές μας συζητήσεις και αποφάσεις για το θέμα του οικολογικού προσανατολισμού. Παρακαλώ κύριε Γέρεπ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Honorable Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω πορίσματα και συμπεράσματα της ειδική ομάδας που εξετάζει το θέμα της βιολογικής προσεγγίσεως όσον αφορά τη γεωργία. Η πράσινη προσέγγιση υιοθετήθηκε το 2013 στη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής σαν μια νέα άμεση πληρωμή που καταβάζει στους αγρότες και ήταν ένας μηχανισμός ώστε να αμείβονται οι γεωργοί για τα αγαθά παράγων και να βελτιωθεί η επίδοση ή ε, περιβαλλοντική όσον αφορά την ΚΑΠ. 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ξοδεύει το πασίνισμα Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίπου 30% όλων των άμεσων πληρωμών τη κοινή ενωτική πολιτική, 8% όλων του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οι γεωργοί πήραν τι πρώτε πληρωμέ του στο πρασίνισμα 100 2016 για αξιώσει που υπευλήθησαν το 2015 Βασικό μας συμπέρασμα από τον έλεγχο είναι το εξής. Το πρασίνισμα έχει εφαρμοστεί. Είναι απίθανο να αυξήσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές επιδόσεις της ΚΑΠ. Οι απαιτήσει περί δεν είναι πολύ απαιτητικέ και ότι αντικατοπτρίζουν κανονικέ αγροτικέ πρακτικέ Λόγω πολλών εξαιρέσεων, οι περισσότεροι γεωργοί, δηλαδή 65% από αυτού, μπορούν να αφεληθούν από μια πληρωμή πρασινίσματο χωρί να υπόκειται σε οδήποτε υποχρέωση στον αυτό το πρασίνισμα τη καλλιέργεια. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το πρασίνισμα οδηγεί σε θετική αλλαγή όσον αφορά τι γεωργικέ πρακτικέ σε πολύ περιορισμένη ε, κλίμακα, δηλαδή 5% περίπου των καλλιεργουμένων γεών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Να σχολιάσω τώρα του αριθμού που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν αποτελέσματα και σαν δείκτε δηλαδή 73-77% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν τουλάχιστον ε, μία υποχρέωση για πρασίνισμα. Ακόμα και αν η εκμετάλλευση έπρεπε να υποχρεώσει την ποικιλομορφία στον άφρα καλλιέργεια και να έχει με ψησπορά σε μόνο ένα εκτάριο από τα 100 εκτάρια η μετρά 100 εκτάρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μέγεθος εκμεταλλεύσεως μετρά κάτω από αυτό το δίκτυο ακόμα και αν δεν υπήρξε καμία αλλαγή όσον αφορά τις πρακτικές της καλλιέργειας διότι ο Γιωργός ήδη σεβόταν τους κανόνες πρασινίσματος ε, πριν επιβληθεί το πρασίνισμα. Αυτός ο δείκτης δεν θα αλλάξει ακόμα και αν υποχρεώσει σύμφωνα με το πρασίνισμα αλλάξουν και σημαντικά εάν παραδείγματο χάρη θα 3, 5, 7% να είναι με πράσινε καλλιέργειε. Λοιπόν, θεωρούμε ότι αυτό ο δείκτη έχει πολύ περιορισμένη χρήση για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τη προσπάθεια βιολογική προσεγγίσεω ή πρασινίσματο. Βρήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θέσει συγκεκριμένου στόχου ή έχει καθορίσει διαφορετικά τι μπορεί να περιμένουμε από το πρασίνισμα, τι θα πετύχει για το περιβάλλον και για το κλίμα περιβαλλοντική και κλιματολογική συνέπεια του πασινίσματος μπορεί να συνδεθεί με, με τη στρατηγική για την προστασία των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ενώσης, για την ποιότητα των εδαφών, που συνδέεται και με τους στόχους για το 2020 Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κλίμα, για την ενέργεια και τους στόχους και το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα του 2030, συμπεριλαμβανόμενο των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου και να συνδέεται επίσης με την βιοπικιλότητα, τη στατική για βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, χωρίς σωστούς όμως στόχους για την ΚΑΠ, δεν μπορεί να υπάρχει μια ολική προσέγγιση για νέε στρατηγικέ συζητήσει για το πρασίνισμα δεν θα πρέπει να στρέφονται γύρω από το θέμα κατά πόσο το πρασίνισμα θα αυξήσει τι περιβαλλοντικέ επιδόσει ή θα μειώσει την επιδείνωση των δικτών των περιβαλλοντολογικών. βλέποντα έναν από του ε, δείκτε, όπω το δείκτη των καλλιεργιών, που ε, μειώθηκε σημαντικά από το 90 μέχρι το 2014. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο, αλλά πόσο θα πρέπει να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ε, ΚΑΠ. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε βασικές, βασικά στοιχεία για βάση των δεδομένων. Λοιπόν, τα κονδύλια για το πρασίνισμα δεν δικαιολογούνται από το περιεχόμενο το περιβαλλοντικό των πολιτικών. Οι πληρωμέ του πρασίνισμα είναι 80 ευρώ κατά εκτάριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξολόγηση συνεπειών θεώρησε ότι το μέσο κόστος για την εφαρμογή των μέτρων του πρασινίσματος δεν θα ξεπερνούσε τα 30 ευρώ και δείχνει η μελέτη διαφορετικό αντίκτυπο για τους καλλιεργητές από λιγότερο από 10% για 40% των καλλιεργητών σε πάνω από 100 ευρώ για 2% των ε, γεωργών. Οι πράσινες πληρωμές παραμένουν ουσιαστικά ένα σύστημα στηρίξης του εισοδήματος Λοιπόν, περιορισμοί σχεδιασμού μειώνουν την αποτελεσματικότητα των τριών πρακτικών που ακολουθούνται για το πασίνισμα. Η ποικιλομορφία των καλλιεργιών δεν θα δώσει πλήρη ωφέλη περιβαλλοντικά για άμυψη σπορά. Χρειάζεται επίσης καλύτερη προσέγγιση για τη μείωση εκπομπών αερίων. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη καλλιεργιών οικολογικών. Χρειάζεται σωστή διαχείριση αλλά δεν είχαμε τα αναμονόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τη βιπικιλότητα. Το πρασίνισμα προσθέτει περίπλοκο χαρακτήρα στην ΚΑΠ. Δεν δικαιολογείται τα αποτελέσματα που αναμένονται από αυτή την προσέγγιση. Η περιπλοκότητα οφείλεται στην αλληλεπικάλυψη μεταξύ πρασινίσματος και άλλων περιβαλλοντικών εργαλείων της ΚΑΠ, όπως ορθή γεωργία και περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μόνη σημαντική διαφορά από ε, την ε, αμοιβή μόρφωση συμμόρφωση είναι ότι κανονικά θα έπρεπε κυρώσει και παραβάσει στο πρασίνισμα να είναι αυστηρότερε. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποίησαν την ευελιξία στην εφαρμογή τη προσεγγίσεω πρασινίσματο, κυρίω όσον αφορά την επιλογή των τυπών ΑΕΦΑ και του καθορισμού των μόνιμων βοσκοτόπων που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι για να βελτιστοποιηθούν ε, τα αποτελέσματα που εφαρμόζονται από τις πολιτικές. Ανταυτού προσπάθησαν να εφαρμόσουν το πρασίνισμα με έναν τρόπο που ελαχιστοποιεί το βάρος για τους καλλιεργητές και για τις χώρες. Βάσει λοιπόν αυτών των πορισμάτων κάνουμε τις εξής συστάσεις για την επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια πλήρη λογική παρέμβαση για τη συνεισφορά της ΚΑΠ σε περιβαλλοντικούς και κλιματολογικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να ακολουθήσει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες οι γεωργοί μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πληρωμές της ΚΑΠ εάν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά κριτήρια και προδιαγραφές που καλύπτονται από τα προγράμματά μας. Χρειάζονται τοπικές ανάγκες, περιβαλλοντικές ανάγκες μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και θα αμείβονται οι γεωργοί για υπηρεσίες που παρέχουν που ξεπερνούν τα ελάχιστα για το περιβάλλον. Τα κάτι μελη θα πρέπει να αποδεικνύουν πριν την εφαρμογή των μέτρων ότι έχουν διαλέξει επιλογές που είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές για την επιτυχία των διαφόρων στόχων που έχουν τεθεί. Κλείνοντα, να πω ποια είναι η ανεπίσημη αξιολόγηση ότι οι αλλαγέ στην τελευταία νομοθεσία Omnibus θα επιφέρει κάποιε βελτιώσει, γι' αυτό τι καλωσορίζουμε. Αλλά βασικά θέματα που αφορούν την απλούστευση και καλύτερε επιδόσει του πρασινίσματο είναι θέματα που πρέπει να επιληθούν στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Αν έχετε τυχόν ερωτήσει, μπορώ να απαντήσω. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γέρεπ, για την πολύ έκθεση και περιεκτική παρουσίαση που μας κάνετε. Το λόγο ζήτησε πρώτα η κυρία Ράνς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γέρεπ από το ελεκτικό συνέδριο που ήρθε στη συνεδρίαση για να μας παρουσιάσει την έκθεση και πραγματικά με εξέπληξαν κάποιες διαπιστώσεις. Δεν με εξέπληξε το 71% των γεωργών ε, δεν εφαρμόζει το, τον οικολογικό προσανατολισμό, γιατί ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων από τους πυλώνες της ΚΑΠ είναι προβληματική. Ε, γι' αυτό επικρίνουμε αυτή την κατανομή των κονδυλίων. Γιατί ουσιαστικά οι μεγαλοκτηματίες καρπώνονται το μεγαλύτερο τμήμα των ενισχύσεων. Το 75% όμω επηρεάζονται από τον οικολογικό προσανατολισμό και αυτό θα πρέπει να το εξάρουμε και να το τονίσουμε. Περισσότερο το ποσοστό της ε, έκτασης που εμπίπτει στον greening είναι σημαντικό, όχι τόσο το ποσοστό των ε, αγροτών που το χρησιμοποιούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας μιλήσατε για το ρόλο της οικολογικοποίησης που θεωρώ ότι είναι πολύ θετικός γιατί ο ρόλος της οικολογικοποίησης του greening είναι το να αναχαιτήσει κάπως την εντατική γεωργία που είναι σαφής πια τάση της γεωργίας λόγω της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Αυτή η οικολογικοποίηση όμως που εφαρμόζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη γιατί είναι και σπάνια σε διεθνές επίπεδο όταν η κυρίαρχη τάση είναι η εντατικοποίηση. Αυτές τώρα οι ενισχύσεις, ε, οι πράσινες, δεν κόστησαν τόσα πολλά χρήματα ε, γιατί η αύξηση των δαπανών ήταν μόνο το 1% λόγω των νέων ενισχύσεων με δεδομένο το τεράστιο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα. Δεν θεωρώ ότι είναι σημαντική αύξηση όπως μας λέτε, αν είναι μόνο 1% των δαπανών για τις ειδικές αυτές οικολογικές ενισχύσεις. Επίσης λέτε ότι όλες οι ενισχύσεις εξαρτώνται από την υλοποίηση των ε, ε, στόχων του περιβάλλοντος. Έτσι όμως στερούμε ε, από τους γεωργούς την ανταγωνιστικότητά τους και μάλιστα σε ένα πλαίσιο που σε συμφωνίες εμπορικέ με τρίτες χώρε. δεν έχουμε αντίστοιχε απαιτήσει από του δικού του γεωργού και έτσι υπονομεύουμε τη δική μα ανταγωνιστικότητα. Οπότε διαφωνώ με αυτή τη διαπίστωσή σα. Και εν ώψη τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική καλό θα ήταν να προσαρμόζουμε την ευρωπαϊκή γεωργία στι ε, περιβαλλοντικέ και κλιματικέ προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του κόσμου ολόκληρου, στο μέτρο όμω που τα μέτρα που απαιτούμε ε, λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, διαφορετικών καλλιεργιών, γιατί έχουμε ε, μόνιμες καλλιέργειες που για προφανείς λόγους εξαιρούνται από, τα, από τις απαιτήσεις της οικολογικής αιρεσιμότητας της τελευταίας ΚΑΠ. Αλλά αν ε, εξαιρέσουμε τους μόνιμους βοσκοτόπους ε, που τόσο πολύ προσπάθεια μας κόστησαν και το προσπαθήσαμε και στο Omnibus. Γι' αυτό είμαστε υπέρ μια αποκέντρωση, μιας περιφερειοποίησης ε, της ε, γεωργικής πολιτικής που κρίνουμε απαραίτητη. Ο κύριο Χόισλινγκ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Μας ξεκαθαρίζουν ότι ουσιαστικά ήταν ε, ένα ξέπλυμα πράσινο και όχι ένας πραγματικός πράσινος προσανατολισμός χωρίς ιδιαίτερη επίδραση για το περιβάλλον. Χαίρομαι για τα στοιχεία αυτά που μας παρουσιάσατε σε ό,τι αφορά το 50% των εκτάσεων που υπάγονται στον πράσινο προσανατολισμό και τελικά δεν ήταν αντίστοιχο το ποσοστό. Θα έπρεπε να μας πει με ειλικρίνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε. Είπατε ότι οι πληρωμές δεν έχουν περιβαλλοντική απόδοση. Δεν έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε, φαντάζομαι, τι θα γίνει στην επόμενη αγροτική μεταρρύθμιση. Πώς μπορούμε να πετύχουμε πραγματική απόδοση και επίδοση. Γιατί είναι το διαρκέ ε, επιχείρημα που χρησιμοποιούμε. Περιβαλλοντική επίδραση και περιβαλλοντική επίδραση. Και τελικά δεν υπάρχει αυτή η απόδοση. Θα πρέπει να απαιτήσουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η απόδοση όταν καλούμαστε να την πληρώσουμε. Ήμουν στις διαπραγματεύσεις και ξέρω πόσοι εργάστηκαν. για να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις προτάσεις του Επιτρόπου τότε. Είπατε ότι εφαρμόστηκε ευελιξία για να μειωθούν τα πρότυπα. Αυτό διαπιστώνουμε και στα κράτη-μέλη. Οι απαντήσεις, ε, η απόκριση στο πράσινο προσανατολισμό είναι πολύ αδύναμη. Δεν είναι δυνατόν να, να περάσει κάτι τέτοιο. Λέει ο Επίτροπος ότι θέλουμε να καταργήσουμε το πρασίνισμα το greening. Λέει δηλαδή ότι είναι πολύ γραφειοκρατικό. Αν θέλουμε όμως κάτι να πετύχουμε στην επόμενη αγροτική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος και θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε και τι ξοδεύουμε για το περιβάλλον. Όχι λοιπόν λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, περιβαλλοντική απόδοση, αλλά πιο πολλά χρήματα για πραγματική απόδοση. Άρα τα χρήματα, οι πόροι θα πρέπει να δεσμευτούν σε επιδόσεις και όχι σε αγροτική έκταση. Να υπάρχει πραγματική πρόθεση περιβαλλοντικής επίδρασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση που μας κάνετε και για την έκθεση. Είσαστε σαφέστατος μετά από ένα χρόνο. Ε, φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε την ψευδέστηση ότι θα αλλάξουν τα πράγματα από μόνο του το επόμενο χρόνο. Θα πρέπει να τα διορθώσουμε τα πράγματα. Αναφέρεται το Omnibus. Θα το αναφέρει και ο κύριος ε, Ντες, ε, βέβαια. Δεν ξέρω τι καταφέρνουμε με το Omnibus. Θα μπορούσαμε να έχουμε ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, δεν το κάναμε και χάσαμε την ευκαιρία αυτή. Ακριβώς εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε να μην υπάρξει περαιτέρω αποδυνάμωση, αλλά ενίσχυση των επιδόσεων των περιβαλλοντικών. Ευχαριστώ κύριε Ντενανό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στην έκθεσή σας επιμένετε ότι η ποικιλομορφία των καλλιεργιών δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά και είναι λιγότερο αποτελεσματική από την αμυσισφορά. Εκεί περιορίζεται η εξάντληση των ε, διαφόρων θρεπτικών σιών του εδάφους και την διάδοση των διάφορων ποθογόνων σιών. Αναφέρεται στη σελίδα 32 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι μια απέτηση για τα φυτά ε, θα μπορούσε να βελτιώσει τα ωφέλη στα, στα όσπρια, ότι αυτή η ιδέα όμω τελικά δεν εφαρμόστηκε διότι υπήρχαν ερωτηματικά όσον αφορά την υποχρέωση συμμόρφωση με τι κανόνε του ΠΟΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό κατά την άποψή μου, διότι οι συμφωνίε ε, είναι πιο προσαρμοσμένε και δεν θα έπρεπε να εμποδίζουν να έχουμε μια στρατηγική που θα ήταν φιλόδοξη και συνεκτική. Λοιπόν, αυτά τα, τα, φυτά που απορροφούν το άζωτο θα πρέπει να καλλιεργούνται ε, σε διάφορα εδάφη και όχι μόνο καλλιέργειες. Τι θα κάνετε το, το θέμα της αμεψισποράς και κυρίως με πρωτενίουχα φυτά που σταθεροποιούν το άζωτο να καλύπτονται τη νέα ΚΑΠ παρόλο που θέλουμε ότι αυτό συνεπάγεται πολύ, πολλά μέσα ελέγχου. Αναφέρατε σαφώς ότι η πρόταση αρχική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρασίνισμα ήταν πολύ πιο φιλόδοξη αυτή που, από αυτή που εθετήθηκε, κυρίως όσον αφορά την επιρροή των 100 μελών και συνεπώς ότι αυτά τα μέτρα που αντιπροσωπεύουν το 30% των αμέσων πληρωμών δεν έχουν δώσει τα κίνητρα που μετρούσαμε. Όσον αφορά το πρασίνισμα, τα κρατη μέλη διαθέτουν ήδη μεγάλο περιθώριο λιγμών, κυρίως όσον αφορά την επιλογή των διαφόρων οικολογικών ε, Χρειάζεται μια νέα ευελιξία που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή ε, πιστεύετε ότι αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία του οικολογικού προσανατολισμού της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω. Δεν φοβάστε ότι θα αποδυναμωθεί η υπόθεση. Να ξεκινήσω αλλιώ όμω να ευχαριστήσω για την ε, σαφήνεια που, ε, και την, ε, τα, τα ανοιχτά λόγια που λέτε. Όποιο είχε διαβάσει την έκθεση, ήξεραν ήδη αυτά που μας είπατε, αλλά το λέτε ξεκάθαρα, σας ευχαριστούμε και το λέτε και από πλευρά δημοσιονομικής, από πλευρά προπολογισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω, πάντα να είμαστε σοβαροί με τα λεφτά του φορολογούμενου. Φόροι είναι αυτοί. Είπατε ότι τα χρήματα χορηγήθηκαν ε, χωρίς επιβάρυνση για τους αγρότες. Τα πόροι αυτοί δαπανήθηκαν για το υπονομαζόμενο πρασίνισμα, χωρίς ε, να υπάρχει όμως αποτέλεσμα για τη βιοπικιλότητα, για το περιβάλλον και το καθεξής. Άρα τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα περιβαλλοντικό. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Οι πόροι αυτοί όχι μόνο σπαταλήθηκαν χωρίς λόγο, αλλά λείπουν και από άλλους σκοπούς τους οποίους θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Διπλή απώλεια και σπαταλήθηκαν α, και δεν έχουμε πλέον τα χρήματα αυτά για τους οικολογικούς σκοπούς της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχίσετε γιατί τα δημόσια αυτά χρήματα θα πρέπει να τα πανώνται στην Ευρώπη μόνο για δημόσιες ε, δαπάνες, για, δημόσιο, για κοινή ωφέλεια για περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε αμετακίνητοι και θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί ε, κανόνες. Αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι μπορούμε να λαμβάνουμε πόρους για να τηρούμε δηλαδή απλά περιβαλλοντικές διατάξεις. Όχι, για να βελτιώσουμε περαιτέρω πέρα από το όριο που έχουν ορίσει οι νόμοι. Παίρνουμε τα χρήματα, τους πόρους. Και θα ήθελα πραγματικά να σας καλέσω να συνεχίσετε να μιλάτε τόσο ξεκάθαρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι πολίτες εντός και εκτός του γεωργικού κλάδου έχουν δικαίωμα να ξέρουν ποιος παίρνει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για ποιους σκοπούς και εδώ. Δεν έχουμε να εξηγήσουμε για τι σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά. Χρειαζόμαστε σαφήνεια. Γιατί παίρνουν οι Ευρωπαίοι αγρότες χρήματα και πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα. Γιατί είναι όλο και πιο μεγάλη η αγανάκτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί κάποιες ομάδες παίρνουν πόρους, ενώ άλλες δεν παίρνουν. Ενώ και άλλοι θα ήθελαν και θα χρειαζόντουσαν ισοδοματική υποστήριξη για να σταθεροποιήσουν το εισόδημά του. Και γι' αυτό λοιπόν από ό,τι φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι οι άμεσες ενισχύσεις, γιατί δεν πετυχαίνουν το στόχο. Άρα σας παρακαλώ να κατονομάσετε σαφείς στόχους, να συνεχίσετε να μιλάνε, να μιλάτε ξεκάθαρα. Όποιος έψαχνε έβρισκε και πριν τα στοιχεία αυτά, αλλά τώρα νομίζω τα λέτε με πιο ανοιχτό τρόπο και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουλουαζό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την έκθεσή του. Το Ελεκτικό Συνέδριο επέκρινε ανοιχτά αυτή την πολιτική πρασινίσματο τη ΚΑΠ, εκφράζοντα τη θλίψη ότι τα, υπήρχαν, δημιούργησαν περιορισμού στα μέτρα για του γεωργού, αλλά είχαν περιορισμένα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Μόνο 5% των εδαφών των γεωργικών είχαν θετικά αποτελέσματα, όπω γνωρίζετε. Αυτό είναι λίγο. Θα πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γεωργών δεν άλλαξαν τι γεωργικέ πρακτικέ ακριβώς για να είναι επιλέξιμη για τις πράσινες πληρωμέ. Μήπως εκεί θα πρέπει να δούμε ότι αυτή είναι η απόδειξη ότι οι γεωργικές πρακτικές ε, δεν είναι και τόσο αντιπεριβαλλοντικές όσο νομίζαμε. Νομίζω ότι το σύστημα που έχει μεταρρυθμιστεί όπω η ΚΑΠ ε, θυσιάστηκαν ούτω ε, διάφοροι γεωργοί που μένουν εκτό του μηχανισμού. θα ήθελα να ξέρω αν οι γεωργοί θα μπορέσουν να βρουν μια υλοποίηση των προσδοκιών τους μέσω της πολιτικής του πρασινίσματος που εφαρμόζονται. Ε, Ευχαριστώ κύριε Νταντά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι αρκετά από την έκθεση που μας παρουσιάστηκε και από το περιεχόμενό της Προσπάθησα εις Μάτιν, δεν βρήκα, πότε συνετάχθη, ποια περίοδο καλύπτει ανάλυση. Όσον αφορά το περιβάλλον, όλοι γνωρίζουμε ότι από, την, από τις πράξεις μέχρι την αντίδραση του φυσικού κόσμου έχουμε μακρά περίοδο, κυρίως ανάλογα με τον τύπο της ε, παρέμβασης με τη επικοινοτητα χρειαστηκαμε χρειαστήκαμε 4-5 χρόνια πριν τα αποτελέσματα της ποικιλομορφία ε, της χλωρίδας να είναι προσμετρήσιμη ε, και να συναρτάται με την πρακτική. Τέλος του 2013 αποφασίσαμε τη μεταρρύθμιση, τέλος του 2013 και σε περισσότερες χώρες μέλη αυτά τα μέτρα ε, τέθησαν μόλις το 2015 σε εφαρμογή. Η Γεωργή είναι επικεφαλής ε, της οικονομικής αυτής προσεγγίσεως ε, και εξελίσσονται οι εκμεταλλεύσεις τους ε, προοδευτικά και αλλάζουν. Αν η έκθεση αναφέρεται στο έτος 2016, πρόκειται περί του δευτέρου έτους εφαρμογής της ε, ΚΑΠ, τον έχουμε 5% των εδαφών που ήδη άλλαξαν καθεστώς, εφαρμόζοντας πρακτικές που συμμορφώνονται περισσότερο με την προστασία των πόρων, αυτό ήδη είναι σημαντικό βήμα. 5% από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια αντιπροσωπεύει σημαντικές ε, εκτάσεις. Εκεί όπου συμφωνώ με το ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά τον ορισμό του στόχου. Ε, πιστεύω ότι αν ήμασταν σαφείς όταν κάναμε τα ρύθμιση όσον αφορά τους προς επίτευξη στόχους, ήταν δύσκολο να περάσουμε από τις μεγάλες ομιλίες και τις θεωρίες στην πράξη. Σε κάποια ερωτήματα τίθενται στα, στους ε, ε, τεχνικούς θεσμούς όσον αφορά τα μέτρα, τα σκόπιμα πρέπει να εφαρμοστούν για να συγκρατείται ο άνθρακας στο έδαφος, να προστατεύονται τα εδάφη, ε, να βελτιώνεται ο αντίκτυπος που έχει η γεωργία όσον αφορά το κλίμα και σήμερα τις πληροφορίες που διαθέτω στις περισσότερες χώρες η γνωστοποίηση αυτών των μεθόδων δεν είναι επαρκής ακόμα. Δεν έχει διαδοθεί στους αγρότες σε μεγάλη κλίμακα. Αυτή η πτυχή μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους γεωργούς έχει μεγάλα, δεν αναφέρεται στην έκθεση. Η κοινή αγροτική πολιτική, πρώτα απ' όλα μια πολιτική οικονομική. Ε, μια πολιτική που στοχεύει καταρχάς στην αντιστάθμιση του γεγονός ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν πληρώνει στο πραγματικό κόστος τη διατροφή του και οι Ευρωπαίοι γεωργοί, συνεπώς όπως οι περισσότερες χώρες του κόσμου, είναι παραγωγή ενός τροφίμου του οποίου μόνο εν μέρη ελέγχουν το κόστος και ότι η δημόσια ενίσχυση είναι εκεί για να τους διασφαλίζει ένα βασικό εισόδημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριος Δεκάστρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ τον Σύμβουλο Γέρεμπ για αυτή τη σημαντική παρουσίαση που μας θέτει διάφορες πτυχές που επανειλημμένα συζητήσαμε στην Επιτροπή μας. Το είχαμε φανταστεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι στον κανονισμό Omnibus θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να πετύχουμε κάποιες αλλαγές. Χαίρομαι που αναφερθήκατε θετικά στις προσπάθειες που κατέβαλε αυτή η Επιτροπή εκμεταλλευόμενη τον κανονισμό Omnibus. Το βασικό στοιχείο, το κεντρικό σημείο είναι η επιλογή ε, μεταξύ τριών μέτρων, τριών μέτρων ποικιλομορφία αμυψισφορά ε, και ε, των τριών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα τα μέτρα και άξονε αυτέ σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε διαφορετικέ φυσικέ συνθήκε. Αν πάμε από τη, από τη Σουηδία στην Κύπρο, πρέπει να εντοπίσουμε μέτρα οικολογικά τα οποία να προσαρμόζονται καλύτερα στι συνθήκε, τι αντικειμενικέ που επικρατούν στη συγκεκριμένη χώρα που εφαρμόζονται. Αυτό μας άρεσε, αυτό που ενέκρινε αυτή η Επιτροπή σε μια έκθεση προηγηθήσα της μεταρρυθμίσεως της ΚΑΠ, όπου λέγαμε ας κάνουμε ένα μενού προτάσεων όπου κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να επιλέγει βάσει των αντικειμενικών συνθήκων που κρατούν βέβαια να είναι υποχρεωμένο να κάνει κάποια πράγματα, ένα αριθμό πραγμάτων, να πετύχει κάποιους στόχους. Αυτή η ευελιξία σίγουρα θα έκανε την ψησφορά ε, να χρησιμοποιείται στη θέση της ποικιλομορφίας ε, ή θα επιλεγόταν άλλες δράσεις σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη μεταρρύθμιση μήπως εκ των πραγμάτων ίσως θα αναγκαζόταν να εφαρμόσει 27 ή 100 γεωρικές πολιτικές και να αφήσει πλήρη ελευθερία επιλογή στα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω. Θα έπρεπε να, να έχει ένα πλαίσιο γενικό και από εκεί τα κράτη-μέλη να επιλέγουν το γενικό πλαίσιο ανάλογα με τα φυσικά αντικειμενικά του χαρακτηριστικά, τι μπορούν να εφαρμόσουν. Ποια είναι η άποψή σα ω ελεγκτικό συνέδριο πάνω σε αυτό. Γενικό πλαίσιο και τα κράτη-μέλη να επιλέγουν λύσει. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και για την παρουσίαση τη έκθεση, ε, διαβάζοντα λοιπόν την έκθεση αυτή διαπιστώνω ότι από ό,τι φαίνεται το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν έχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. Κοιτάζοντα τι εκτάσει στη Γερμανία. Έχουμε 20.000 ε, ε, εκτάρια ανά για ε, αναδίκηση. Έχουμε εκτάρια για παγίδευση άνθρακα, για βιοπικιλότητα και έχουμε και κάποιες μικρότερες εκτάσεις. Αυτά λοιπόν δεν λαμβάνονται υπόψη. Ένα τρίτο των εκτάσεων στη Γερμανία ήδη συμμετέχει σε θελούσιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες διτάξεις και να προσθέσουμε γιατί ήδη ισχύουν. Και επίσης ε, αυτό που με εκνευρίζει είναι το πώς ε, εκτιμά το και υπολογίζει το ελεκτικό συνέδριο τις ενδιάμεσες ε, καλλιεργίες. όπου υπάρχει συλλογή των καρπών το φθινόπωρο και ε, χρησιμοποιούνται για τα βιοκαύσιμα. Πλέον αυτές οι ενδιάμεσες καλλιέργειες ε, ε, παραμένουν και στην άνοιξη όμως όταν πλέον συλλέγονται οι καρποί δεν έχουν τόσο μεγάλη απόδοση όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έχετε λάβει υπόψη. Πώς να θεωρήσω λοιπόν ότι είναι από τεχνικής άποψης άρτια αυτή η έκθεση. Πολύ λυπάμαι, αλλά Νομίζω ότι οι, οι υπάλληλοι του εκτικού συνεδρίου θα πρέπει να έχουν μισθό μόνο εφόσον έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Και αυτή την εμπειρογνωμοσύνη ειλικρινά δεν τη βλέπω στην έκθεση αυτή. Κύριε Φλάνναγκαν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έλαβα την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού χτες και συμμετείχα στη συζήτηση και να σα πω ότι ήταν εντελώ διαφορετική η ατμόσφαιρα χθε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού σε σχέση με σήμερα. Λε και ζούμε στην Επιτροπή με αυτή σε μια φούσκα. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέγεται. Εκτό τη επιτροπή μα. άκουσα ένα μέλο να λέει μόνο ένα μόνο βουλευτή ότι δεν κοστίζει πολύ. Ε, 8% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Σε καιρούς ε, συνολικών συζητήσεων για όλο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη και του Brexit και μετά από τα έγγραφα συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, προσπαθώντα να αποφασίσουμε τι ποσοστό του προπολογισμού θα συνεχίσει να δαπανάτε στην Γεωργία. Αν ήσασταν λοιπόν χθε στην συνεδρίαση τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, θα βλέπατε ότι προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να διατηρήσουμε το 8%. Εγώ θα προσπαθήσω μέχρι τελευταία ε, πτώσεω, αλλά... Αυτά που συμβαίνουν δεν μας δυσκολύνουν τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου βλέπουμε το ελεκτικό συνέδριο από δική μου εμπειρία θεωρώ ότι αποτελεί ένα θερμόμετρο. Το θερμόμετρο υποδεικνύει τη θερμοκρασία και σήμερα τι μας λένε, ότι δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα του θερμομέτρου. Δεν δουλεύει το θερμόμετρο και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε γιατί δεν έχει πρόβλημα η θερμοκρασία μας είναι λυπηρό, το ξέρω, λέει η πραγματικότητα είναι διαφορετική γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί ο φορολογούμενος στην Ευρώπη εκτός και οι βουλευτές, αν θέλετε, εκτός της Επιτροπής μας, δεν είναι τόσο ήσυχοι ότι όλα πάνε καλά. Και θα πρέπει να, προσω... προστατεύσουμε τον, προϋπολογισμό τον προπολογισμό μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να δαπανώνται σωστά οι πόροι. Μιλάμε λοιπόν για τις χώρες και για τις επιλογές που έχουν οι χώρες. Οι επιλογές που είχε η Ιρλανδία σε πολλές περιπτώσεις. Ο κόσμος που ήδη λάμβανε μεγάλες πληρωμές, μεγάλες ενισχύσεις, έλαβε ακόμα πιο μεγάλες ενισχύσεις για το πρασινίσμα. Και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές. Αυτό προφανώς είναι μεγάλο πρόβλημα. Διαφορές ανά έκταση και ανά ε, εισόδημα. Και έχω παραπονεθεί και στο παρελθόν για την έλλειψη συμμετοχής βουλευτών εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί έχω ακούσει πολλούς βουλευτές να χύνουν κροκοδίλια άκρια για τις απώλειες στη γενικό προπολογισμό. Αν με τους ένοιαζε και τους έκοπτε, πού είναι σήμερα και φαντάζομαι ότι στην παρούσα φάση κάθονται και γράφουν ανακοινώσει τύπου για το πώ τρομερό θα ήταν αν υπήρχαν μειώσει τον προπολογισμό για τη γεωργία. δεν είναι όμω εδώ να τον προασπιστούν. Ο πρόεδρο. Ε, σίγουρα. δεν καθορίστηκαν οι ζώνες οικολογικής εστίασης ε, στις, στους, ε, στα ίδια μέρη που είχαμε και, τους, ε, και τις ενισχύσεις για να στηριχθεί το γεωργικό εισόδημα και να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα. Αν ήταν αποτυχημένος ο τρόπος ε, οικολογικής, ε, οικολογικής προσανα, οικολογικού προσανατολισμού, τότε θα πρέπει ε, να δούμε τι έγινε με τις ενισχύσεις. Ίσως οι ενισχύσεις της οικολογικοποίησης ε, περισσότερο ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα και το αγροτικό εισόδημα παρά τον οικολογικό προσανατολισμό. Αυτό θα πρέπει να το αναρωτηθούμε. Ο κύριος Μπογκόβιτς. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον κύριο ε, Γιάρεπ από το ελεκτικό συνέδριο που ήρθε και να μας παρουσιάσει την έκθεση και τον ευχαριστώ ε, για, το, για τη δύσκολη αυτή έκθεση που εκπώνησε το ελεκτικό συνέδριο που για να την ε, συντάξει χρειάστηκε να αξιολογήσει την εφαρμογή των στόχων από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και διαπιστώνουμε ότι η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου καταδεικνύει τις δικές μας ουσιαστικά ελλείψεις και αδυναμίες, γιατί δεν προσδιορίσαμε παρκώς την πολιτική και τους στόχους του οικολογικού προσανατολισμού. Οπότε Τα κονδύλια της γεωργίας υποτίθεται θα μας εξασφαλίσουν ε, ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα, ε, υγιεινό αέρα να αναπνέουμε, πλούσια εδάφη, αλλά ο γεωργικός ε, προϋπολογισμός όλο και συρρυκνώνεται. Επίσης, εξετάζοντας τα γεωργικά εισοδήματα, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα από τα εισοδήματα άλλων κλάδων παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ώστε και η γεωργία να είναι πιο προσοδοφόρα γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Επίσης διαπιστώνουμε ότι το 30% των κονδυλίων είχαν προβλεφθεί για τις άμεσες ενισχύσεις και εδώ μιλούμε για ένα σύστημα που θα επηρεάσει το σύνολο της Γεωργίας. Διαρωτόμαστε λοιπόν αν οι στόχοι που θέσαμε είναι σωστοί και αν όντως θα εξασφαλίσουν πιο ποιοτικά τρόφιμα, καθαρότερο αέρα και πιο παρα... εδάφη. Θα πρέπει η γεωργία να σέβεται ταυτόχρονα το περιβάλλον και να αποτρέπει τη, τις κλιματικές αλλαγές. Δεν πρόκειται όμως το 5% των άμεσων ενισχύσεων να το δώσουμε στο 10% ε, της ε, αγροτικής γης που θα παράγει μόνο το 2% των τροφίμων. Δεν είναι λογικό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στον προσδιορισμό της νέας πολιτικής και των στόχων μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι επιδιώκουμε και να μην ξεχνούμε ότι καλύπτουμε περίπου το 75-80% της, ε, των γεωργικών εκτάσεων. Και το 5% αφορά συγκεκριμένες ε, γεωργικές και συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές ε, φιλοπεριβαλλοντικές, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο αρνητική εντύπωση που έδωσε η έκθεση, απλώς επισημαίνει την ανάγκη να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τους μελλοντικούς μας στόχους και αυτή είναι σημαντική πρόκληση γιατί στο μέλλον θα έχουμε πολύ λιγότερα χρήματα ανά εκτάριο στο διαθέσιμο γεωργικό προϋπολογισμό. Και επίση θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για την ηλικιακή ανανέωση, για να προσελκύσουμε και νέου στη γεωργία. Γιατί θέλουμε αύξηση του αριθμού των γεωργών που θα εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που θα είναι οικολογικές, φιλοπεριβαλλοντικές και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε κάποια χρήματα στα μέτρα αυτά, γιατί μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε τη γεωργία μας και θα προστατεύσουμε ταυτόχρονα και το περιβάλλον μας. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σωστά αυτό που είπε ο Μισελ Νταντών, ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι δύσκολα επιτεύχθουν σε δύο-τρία χρόνια. Επίση αληθεύει τα μέλη τη Παρού Επιτροπή δεν ήταν ικανοποιημένοι με τι προτάσει περί οικολογικής προσεγγίσεω που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη τελευταία μεταρρύθμιση. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τα μέτρα. Τι μα έλειψε. Ήταν μια κίνηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει στον πυλώνα ένα τα αποτελέσματα περιβαλλοντικά. Αυτό ήταν ο στόχο κατά την απόψή μου και αυτό επετεύχθη. Και ίσως μπορείτε να το σχολιάσετε. Δεν υπάρχει σύγκρουση στα συμπεράσματά σας και πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο στήριξη του εισοδήματο το πρασίνισμα. Οι πληρωμές του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ αυτό αφορούσαν. Τα χωρίσαμε σε δύο τμήματα, αλλά ήταν τα ίδια χρήματα και σαφώς οι γεωργοί δεν κάνουν αυτή τη διάκριση. Αυτό που λέγουν είναι ότι αυτό υποστηρίζει το εισόδημά μου. Και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, των οποίων την άποψη ξέρω, γιατί γνωρίζω πολλούς, λέω ότι πρέπει να δουν το μέσο εισόδημα ε, της γεωργίας στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μεγάλες πληρωμές και αυτό πρέπει να αλλάξει. Κοιτάξτε όμως το μέσο όρων το μέσο όρο πρέπει να κοιτάμε όταν λαμβάνουμε αποφάσεις, όχι τις μεγάλες πληρωμές που βγαίνουν στους τίτλους των εφημερίδων, διότι υπάρχουν συνέπειες αν δεν προστατεύσουμε τον προπολογισμό. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη, το ελεκτικό συνέδριο αναλύει τώρα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική μορφή της ΚΑΠ. Έχω ανησυχίες πραγματικές όσον αφορά τα διάφορα σημεία που αναφέρεται εκεί για το μέλλον, της προτάσει σα για το μέλλον της ΚΑΠ. Διότι αν ποτέ την απλούστευση και τις προτάσεις σας τις βάζουμε μαζί δεν θα λειτουργήσουν. Διότι αυτό που προτείνεται είναι απίστευτα περίπλοκο σαν ιδέα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει. Και ειλικρινά ανησυχώ διότι σε πολλά κάτι μέλη συμπεριλαμβανομένου του δικού μου τι βλέπουμε ότι πολύ καλοί ε, βιότοποι στις ε, εκμεταλλεύσεις εξαλείφονται για να πει ένας βιότοπος για να ενταχθεί σε νέο σχήμα που έχει σχεδιάσει η Ευρώπη το κάτω μέλος. Ενώ αν πληρούσαμε για τους, παρούς, τους παρόντες βιοτόπους δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Βλέποντας την έκθεσή σας αυτό δεν αρκεί. Δεν θέλετε να μήψετε τους γεωργούς για την παρούσα συνεισφορά τους στους περιβαλλοντικούς στόχους. Χαίρομαι που κουνά το κεφάλι σας διότι διάβασα ξεκάθαρα αυτό που λέω. Και πρέπει να λέτε σαφέστατα ότι η μεγάλη βλάβη που κάναμε στην Ευρώπη ποια είναι. Δεν επιτρέψαμε σε φυσικές περιοχές της εκμεταλλεύσεις να αμυφθούν στην ΚΑΠ. Και ίσως προχωρώντας προς το μέλλον πρέπει πρώτα αυτό το θέμα να καλύψουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαγκίνες. Σίγουρα εστερνίζομαι τις απόψεις και τις αξιολογήσεις που κάνατε για την οικολογικοποίηση και την διατήρηση κάποιων τέτοιων οικοτόπων. Ο κύριος Ροπέ, σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γενικώ έχω πολλές συναντήσεις με Γιώργους και δια... Πιστώνω ότι το ζήτημα της οικολογικοποίησης είναι ένα επίμαχο θέμα και επώδυνο για αυτούς. Και χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσει το πρόβλημα. Μερικοί είχαν πολύ ψηλέ προσδοκίες, άλλοι πολύ λίγες. Και εσείς είπατε τελικά ότι ο κόσμος, οι αγρότες δεν εισέπραξαν αυτό που περίμεναν. Και το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί δεν αρκεί και ούτε ο περιβαλλοντικός το αντίκτυπος είναι σημαντικός. Αλλά από τη στιγμή που ο Γιώργος δεν έκανε αυτά που έπρεπε, δεν θα λάβανε τις ε, ενισχύσεις. Αλλά ακόμη και αν πληρούσε τις προϋποθέσεις, μερικές φορές ε, ε, και πάλι δεν μέναμε ικανοποιημένοι ή μερικές φορές τα κριτήρια ήταν πολύ αυστηρά. Και δεν ξέρω γιατί καταλήξατε τελικά σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί ήδη στη συζήτηση είπαμε ότι μια πολύ σημαντική πτυχή του πρασινίσματος είναι ότι ε, χάρη σε αυτό οι αγρότες είχαν συμπληρωματικές δραστηριότητες και επιπλέον κόστος χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνουν ε, επιπλέον εισόδημα τα κονδύλια που υπήρχαν διαθέσιμα στο παρελθόν απλώς ανακατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Ενώ από τη στιγμή που έχει υψηλότερο κόστος ο Γιώργος θέλει και περισσότερα χρήματα, αύξηση του εισοδήματος. Οπότε, αν προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα θα πρέπει να το τροφοδοτούμε με νέα κονδύλια. Γιατί αλλιώ το κόστος για το Γιώργο αυξάνεται, οι ζημίες αυξάνονται, το, αυξάνονται, το κέρδος μειώνεται και η γεωργία που ούτως ή άλλως δεν είναι ελκυστική απασχόληση λόγω της κρίσης, θα γίνει στο μέλλον ακόμη λιγότερο ελκυστική. Γιατί είναι πολύ χαμηλό το γεωργικό εισόδημα και αν δεν αποζημιώνουμε τους γεωργούς ε, για τις ζημίες τους ή για το κόστος που καταβάλουν, τότε δεν πρόκειται να έχουμε ε, ε, επάρκεια στη γεωργική παραγωγή τροφίμων ή ποιοτικά τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Επίσης, ε, όταν αναθέτουμε σε όλους παρόμοιες υποχρεώσεις, γιατί τα προγράμματα τα, της οικολογικοποίησης ε, είναι παρόμοια, ενώ οι πληρωμές είναι πολύ διαφορετικές, οι ενισχύσεις είναι διαφορετικές. Ένας αγρότης που παίρνει το 50% σε σχέση με αγρότη γειτονική χώρα και παρόλα αυτά έχει τι ίδιε υποχρεώσει. Το θεωρείτε δίκαιο αυτό, ενώ οι υποχρεώσει είναι ίδιε, η ανταμοιβή να είναι πολύ διαφορετική. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αγορετών. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργία. Α, συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Μπούντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα θέλαμε όλοι οι γεωργοί να έχουν ε, επαρκή έσοδα για να μπορούν να ζουν. Να ζουν σωστά και καλά. Και συχνά μας ρωτούν γιατί οι γεωργοί παίρνουν τόσα πολλά χρήματα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι σε τελική ανάλυση οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν και ένα εισόδημα το οποίο να του επιτρέπει να ζουν, να ζουν με αξιοπρέπεια. Στον τομέα τη υπέτρου αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και χρειαζόμαστε και τρόφιμα καλή ποιότητα επιπλέον για όλου του πολίτε ασφαλώ. Έχω επισκεφτεί γεωργού. έχω πάει στο σπίτι του. Όλοι λοιπόν θίγουν το ίδιο θέμα, το θέμα των κυριώσεων. Ότι συχνά δηλαδή γίνονται σφάλματα, λάθη, και τα λάθη αυτά ουσιαστικά οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης από πλευρά των αρχών, ότι δεν είναι σαφές σε τελική ανάλυση το τι θα πρέπει να γίνει και τελικά παραβιάζουν κανόνες χωρίς να γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν οι κανόνες. Τελικά τα, οι κυρώσει είναι πολύ υψηλέ και τελικά τους οδηγούν σε αναστολή των δραστηριοτήτων τους. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο και τους ε, συνεργάτες ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις διαρκείς ε, και σταθερές επιδόσεις και με ενισχύσεις που μας δίνουν. Χαιρόμαστε που συζητάμε λοιπόν αυτή την έκθεση σήμερα και ακούσαμε διάφορους συναδέλφους και πολλά από τα προβλήματα υπογραμμίστηκαν. Κάτι άλλο θεωρώ που θα, θέλουμε, θα θέλαμε να τονίσουμε έχουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, για την οποία λυπούμαστε, και αυτή θα επιφέρει ε, απώλεια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο σε εισφορές. Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της σε, διάφορες, ε, σε τομείς. Σε ό,τι αφορά τα 12 δισεκατομμύρια αυτά φυσικά, σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα δεν μιλάμε για το ίδιο για το ίδιο μέγεθος ε, κλίμακας. Ε. Κάτι άλλο. Ο συνάδελφος ε, δεν έχει, δεν κάνει λάθος όταν λέει ότι δεν είναι δυνατόν τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά να προσμετρούνται και να καταμετρούνται στην αποδοσή τους σε ένα-δύο χρόνια. Είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε λοιπόν από τώρα κατά πόσον κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση γιατί μας λείπει η συνολική εικόνα για την παρέμβαση την οποία προσπαθούμε να πετύχουμε. Δεν έχουμε θέσει και σαφείς στόχους. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι αν δεν υπάρχουν τέτοιοι σαφείς στόχοι και για τη μελλοντική ΚΑΠ, και αυτό προφανώ είναι μια εκτενή διαδικασία, θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Θα είναι πολύ γενική η μέθοδος υπολογισμού, αλλά δεν θα μπορούμε να καταδείξουμε με συγκεκριμένα αποτελέσματα το τι έχουμε πετύχει και τι συνέβη πραγματικά σε ό,τι αφορά με τα πιλωτικά προγράμματα όπως το ΛΙΖΑ. Ε, Ενδεχομένω να είχαμε ένα σημείο αναφορά. Και συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί νομίζω ότι χανόμαστε σε συζητήσεις και βρισκόμαστε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο όπου υπάρχουν και μια σειρά άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα για την βιοπικιλότητα, για το πακέτο για την ενέργεια, για την ε, στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Όλες αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να συνενωθούν και τότε μόνο μπορούμε να είμαι για ένα πραγματικό πράσινο προσανατολισμό. Όχι πράσινη διακόσμηση, πραγματικά οικολογικό προσανατολισμό. Αλλά σε κάποιους τομείς πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι απογοητευμένη σε ό,τι αφορά και τους ε, συναδέλφους που λένε ότι εντάξει, ε, καλά τα κάνουν και οι αγρότες, ό,τι μπορούν να κάνουν και αυτοί και ας συνεχίσουμε στην πεπατημένη. Δεν νομίζω ότι αυτό α, ικανοποιεί τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ο... Οι πόροι αυτοί οι οποίοι κατανέμονται δεν έρχονται από το πουθενά. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει να ξέρουμε τι θα παράτε, για ποιο σκοπό, πού βρίσκεται αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Άρα χρειάζονται αυτοί οι έλεγχοι. Αν λοιπόν δεν έχει το ελεκτικό συνέδριο τη δυνατότητα εξαγωγη των ελέγχων, γιατί δεν έχει τι αντίστοιχε παραμέτρου, εμεί ε, πώ θα τα δικαιολογήσουμε όλα αυτά στου φορολογούμενου και τότε ανακύπτουν οι συζητήσεις σαν αυτή που έγιναν εν ώψη του επόμενου που Αν δεν έχουμε λοιπόν τα δεδομένα, αριθμητικά στοιχεία, με τα οποία να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτά οι πόροι, public, ε, τα δημόσιοι πόροι, να παρούνται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντό και ότι επιδεικνύουμε αλληλεγγύη για την επίτευξη ε, ευρωπαϊκών στόχων, δεν θα έχουμε σωστή συζήτηση. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνση Γεωργία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Πιέρ Μπασκό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που έχουμε ανταλλάξουμε απόψεις για την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου περί του πρασινίσματος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τη Γεωργία, για την παρούσα ΚΑΠ και για τη μελλοντική ΚΑΠ. Καταρχά να υπογραμμίσω κάτι, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει αυτή την ειδική έκθεση και την ουσία όλων των συστάσεων. Την αποδεχόμεθα και θα ληφθούν υπόψη όταν θα οικοδομήσουμε μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική για τη μελλοντική ΚΑΠ. Το συνέδριο εντοπίζει κάποιες αδυναμίες των πρασίνων μέτρων, κυρίως αν αφορά τις επιδόσεις και τον περίπλοκο χαρακτήρα τους. Παραδεχόμαστε πολλά από αυτά που αναφέρονται, παρόλο που κατά την άποψή μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δοθήσεις της χρονικής ειστερήσεως μεταξύ παρεμβάσεως ε, και εφαρμογή πρακτικών και αποτελεσμάτων για τα εδάφη, το νερό, βιοποικιλότητα, κλίμα. Ε, επανειλημμένα ακούστηκε αυτό στη συζήτηση. Όμως, να πω ότι κάποια πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου, κατά την άποψή μας, είναι πολύ σημαντικά προς βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών επιδόσεων της γεωργίας στο μέλλον και πολύ σημαντικά στοιχεία τόσο ώστε να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα, τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Υπενθυμίζει η έκθεση την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρασίνισμα έχει δυνατότητες να βελτιώσει περιβαλλοντικές και κλιματολογικές επιπτώσεις της μελλοντική ΚΑΠ σε σχέση με την ΚΑΠ διότι ε, 77% ε, ε, των καλλιεργουμένων εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες για ε, το πρασίνισμα και πρέπει να δούμε όχι μόνο το ποσοστό των εδαφών, αλλά και το ποσοστό των καλλιεργητών για το περιβάλλον και το κλίμα. Και αυτός ο μέσος όρος συγκρίνεται με το 25% περίπου των αγροτικών ε, περιβαλλοντικών μέτρων που εφαρμόζονται. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο για το περιβάλλον και το κλίμα όσον αφορά την αλλαγή των διαφόρων πρακτικών. Η έκθεση του συνεδρίου δείχνει ότι οι καλλιεργητικέ πρακτικέ επηρεάζονται από τι απαιτήσει περιπρασινίσματο. 13% των εκμεταλλεύσεων που επισκέφθηκε το ελεγκτικό συνέδριο εφάρμοσε πρακτικέ ποικιλομορφία καλλιεργιών και 37% των εκμεταλλεύσεων αλλάζουν τις πρακτικές όσον αφορά την ε, οικολογική προσέγγιση. Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα με την θέσπιση και εισαγωγή του πρασινίσματος ε, στη φάση της εφαρμογής. Θα δούμε μετά ποια είναι τα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Να επιστρέψω και σε μία από τις βασικές επικρίσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που ακούστηκε στη συζήτηση άλλωστε. Επέκρινε το γεγονός ότι οι πράσινες πληρωμές πληρώνουν για πρακτικές που ίσως να εφαρμόζονται ήδη από τους γεωργούς και στην έκθεση θεωρείται σαν απόβαρο, αναφέρεται σαν απόβαρο. Κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρασίνισμα δεν έχει σαν στόχο απαραίτητα τη μεταβολή των πρακτικών των καλλιεργητικών των γεωργών, αλλά να υποστηρίξει την παραγωγή αγαθών που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτή η διευκρίνηση είναι πολύ σημαντική. Να έχουμε υπόψη ότι το πρασίνισμα δεν λειτουργεί σαν αγροπεριβαλλοντικό όπως τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που θέλουν να αποζημιώσουν τους γεωργούς για αλλαγή πρακτικής και είναι σημαντικό εάν οι γεωργοί εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές που θεωρούνται εποφελείς για το περιβάλλον και το κλίμα είναι σημαντικό να μην υπόκειται σε κυρώσει γι' αυτό, να μην βρίσκουν την θέση. Και οι πράσινε πληρωμέ εμποδίζουν να αποφύγουμε την επιδείνωση των πρακτικών. Αναφέρθηκε αυτό το πρωί. Τα τελευταία 30 χρόνια είδαμε μια τάση προς εντατικοποίηση και μονοκαλλιέργειες και είναι σημαντικό και αυτό, συμφωνούμε σε αυτό, με το πρασίνισμα να τα αποφύγουμε αυτά. Να αποφύγουμε συνέχιση της τάσης και να σταματήσει αυτή ε, η επιδείνωση. Σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το ελεκτικό συνέδριο είναι στην έκθεση του 2016 για την πρώτη εφαρμογή του πρασινίσματος ότι η εφαρμογή του πρασινίσματος από τα κράτη-μέλη και από τους γεωργούς των κρατών μελών δεν επέτρεψε την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το πρασινίσματο θα πρέπει να τονιστεί και να αναγνωριστεί και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο χρόνο πρότεινε απλούστευση, εναρμόνιση και βελτίωση κάποιων απαιτήσεων περί πρασινίσματος για να αυξηθούν τα περιβαλλοντικά ωφέλη του πρασινίσματος και αυτή η βελτίωση έχει σαχθεί σαν κατεξισοδότηση κανόνας που θα τεθεί σε ισχύ ε, αρχές ενεστώτος έτος. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Μιλάμε για την τρέχουσα ΚΑΠ και το πασινίσμα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά το 2020. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνη την άποψη του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι σε πολλέ χώρε το πρασίνισμα εισήχθη υπό την παρούσα μορφή σε μια μορφή που είναι πολύ περίπλοκη, πολύ γραφειοκρατική και δεν είναι αρκετά ευέλικτη ούτω ώστε να κατορθώσει να πετύχει τελικά τους στόχους μας περιβαλλοντικούς, τους φιλόδοξους. Και θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Γι' αυτό και πολύ απλούστεροι όσον αφορά το περιβαλλοντικό και το κλιματολογικό μέτωπο στο μέλλον. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφέ την ανακοίνωσή τη που υιοθέτησε τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωση για το μελλοντικό τομέα των τροφίμων και τη καλλιέργεια ε, και η πράσινη αρχιτεκτονική δεν θεωρείται σαν η βέλτιστη ε, αρχιτεκτονική για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις καλύτερες επιδόσεις και περαιτέρω ε, απλούστευση. Γι' αυτό Χρειάζεται μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική που βασίζεται σε θετικέ εμπειρίε που αποκομίσαμε. Είχαμε πολλέ θετικέ εμπειρίε από το πρασίνισμα και τη διασταυρούμενη συμμόρφωση. Θέλουμε να βασιζόμαστε περισσότερο στι επιδόσει και όχι στη συμμόρφωση. Και θα χρησιμοποιούμε πλήρω τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή η νέα προσέγγιση και αυτή η νέα πράσινη αρχιτεκτονική θα αποτελεί ένα τμήμα τη νομοθετική προτάσεω για το μέλλον τη ΚΑΠ που θα υποβληθεί αργότερα φέτος το 2018 και βάσει αυτή τη νέα προσεγγίσεω, τα κράτη-μέλη θα περιγράψουν σε στρατηγικό σχέδιο, όπω το αποκαλούμε, το πώ προτίθενται να πετύχουν περιβαλλοντικού και κλιματολογικού στόχου που θα καθορίζουν τα ίδια βάσει γενικών ευρωπαϊκών στόχων και η αιρεσιμότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη διάφορε πολιτικέ ε, για όλε τι πληρωμέ τη ΚΑΠ και θα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η νέα προσέγγιση, η νέα λογική παρεμβάσεων, η οποία αποτελεί αντικείμενο διεξοδική ανάλυσης και προβληματισμού, τόσο ώστε να μεταμορφωθεί σε μια ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ο του Ενεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας ε, και τα σχόλια που υποβάλλατε. Ε, το κεντρικό θέμα στη συζήτηση είναι οι στόχοι. Και αυτό το συζητήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Ε, ο ελεγκτής δεν πρόκειται να θέσει εκείνο τους στόχους. Με το ισχύον σύστημα το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε σαφείς στόχους. Όπως επισήμανε και ο κύριος Μπόγκοβιτς και άλλοι. Και γι' αυτό τελικά ε, μιλάμε για τα μέτρα που επιλέγονται, αν είναι κατάλληλα και πώς εφαρμόζονται. Αλλά πριν περάσουμε στα μέτρα, πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους στόχους. Και αυτό λένε οι συστάσεις μας, ότι πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους στόχους των μέτρων, αν θα είναι η εισοδηματική στήριξη ή ο οικολογικός προσανατολισμός. Και η ΚΑΠ θα πρέπει να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές ε, και κλιματικές επιδόσεις της κοινής γεωρικής πολιτικής. Αλλά αυτό είναι θέμα νομοθέτη, όχι ελεκτικού συνεδρίου, να καθορίσει τους στόχους. Και εμείς θα ε, ελέγξουμε κατόπιν αν όντως έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι. Χθες ε, ε, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού με το συμπέρασμα ή την εξήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν γίνεται ανακατανομή των ενισχύσεων. Όλοι οι αγρότε λαμβάνουν τι ίδιε ενισχύσει με πριν το greening. Και αν δείτε και την έκθεση, διαπιστώνετε ότι δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα πράγματα στι γεωργικέ πρακτικέ. Οπότε ήταν όντω μεγάλη μεταρρύθμιση της πολιτικής ε, της ΚΑΠ το 2013. Μάλλον όχι. Οπότε ξαναρχόμαστε στο ζήτημα των στόχων του πρασινίσματος και εμείς οι ελεγκτές δεν πρόκειται να θεσπίσουμε τους στόχους, αλλά δεικνύουμε την έλλειψη των στόχων που στο μέλλον θα πρέπει να είναι σαφέστερα προσδιορισμένοι. Ο κύριος Νταντάν ρώτησε ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος μετά από μια πενταετή εφαρμογή και ότι είναι πολύ σύντομος ο χρόνος για να το κρίνουμε. Συμφωνώ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές και διαπιστώσαμε μόνο ότι 5% των Ευρωπαίων αγροτών έκαναν κάποιες αλλαγές. Και ακόμη και σε αυτό το ποσοστό το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο, γιατί ουσιαστικά είναι η επιπλέον προστασία ότι οι μόνιμοι βοσκότοποι δεν θα, δεν οργωθούν, αλλά οι γεωργικές πρακτικές δεν έχουν αλλάξει ε, αισθητά. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε εντυπωσιακό περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή ε, εντυπωσιακή βελτίωση ε, των εκπομπών αερίου του θεροκηπίου εφόσον δεν διαπιστώνουμε αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές. Η κυρία Μαγκίνες είπε ότι δεν αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι θα πρέπει πρέπει να επιβραβευθούν για κάτι που ήδη κάνουν. Αλλά οι αγρότες δεν είναι όλοι στην ίδια θέση. Κάποιοι αγρότες έχουν καλές κατάλληλες πρακτικές, αλλά άλλοι γεωργοί δεν έχουν σωστές πρακτικές. Οι γεωργικές πρακτικές μερικές φορές παρά είναι εντατικέ και βλάπτουν το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε διαφορετικούς στόχους ανάλογα με τα διαφορετικά είδη της γεωργίας και των γεωργικών πρακτικών και να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες ή τις διαφορές των κρατών μελών. Ο κύριος Δεκάστρο ρώτησε τι γίνεται με τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών. Έχουμε, στο μέλλον θα έχουμε 27 διαφορετικές κοινέ γεωργικές πολιτικές. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις και ίσως επιλέγουμε διαφορετικό τρόπο κάποια μέτρα. Και αυτό ισχύει και για τις ε, περιοχές οικολογικής εστίασης της ΕΦΑΣ. Αλλά στο δεύτερο πίνακα, στη σελίδα 37 της έκθεσης, δείξαμε ότι η Πολωνία και η Ολλανδία, για παράδειγμα, έχουν μελετήσει ποιες ε, περιοχές οικολογικής εστίασης είναι οι κατάλληλες για τις δικές τους χώρες. Και παρά όλε τις συστάσεις που έδωσαν οι εμπειρογνώμονες, τελικά οι δύο χώρες δεν ακολούθησαν αυτές τις συστάσεις των ειδικών. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν τα εθνικά προγράμματα των 27 χωρών είναι κατάλληλα και τα επιλεγμένα μέτρα είναι όντως κατάλληλα για να υλοποιήσουν τους στόχους που θα θέσουμε. Η κυρία Μαγκίνες ρώτησε αν θα δημοσιεύσουμε κάποια ανακοίνωση. Ναι, ε, ετοιμάζουμε ένα ενημερωτικό σημείο για το μέλλον της ΚΑΠ που θα εκδοθεί προς τα τέλη Μαρτίου και θα τροφοδοτήσει και αυτό τη συζήτηση για το μέλλον της του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιο, το μελλοντικό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριο Ροπέ ε, ρώτησε αν είναι διαφορετικέ οι ενισχύσεις ε, των αγροτών και αν ε, με διαφορετικές ενισχύσεις καλούνται να υλοποιήσουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Αυτό όμως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το greening, γιατί το greening αφορά τις βασικές ενισχύσεις. Οι βασικές ενισχύσεις είναι διαφορετικές. Το greening όμως, η οικολογικοποίηση είναι συνήθως στα περισσότερα κράτη-μέλη, είναι ένα ποσοστό των βασικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες. Και όπως ξέρετε υπάρχει μια διαδικασία εξομοίωση στο μέλλον των επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων. Επίσης είπατε ότι οι Γεωργοί έκαναν αυτό που περιμέναμε από αυτούς. Και αυτό είναι και το πόρισμα της έκθεσης, ότι τα κράτη-μέλη και οι Γεωργοί αντιμετώπισαν το greening ως μια επιπλέον επιβάρυνση και περιπλοκή και προσπάθησαν να βρουν το, την εύκολη λύση ε, να εξασφαλίσουν τις ε, ενισχύσεις χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες στο greening. Εγώ όμως είπα, αν όντω δεν υπάρχει αλλαγή των γεωργικών πρακτικών και προσπάθεια για να δοθεί οικολογικό προσανατολισμό, όντω το greening θα μείνει ω μια επιπλέον επιβάρηση και περιπλοκότητα τη κοινή γεωργική πολιτική. Και ένα από του στόχου τη νέα ΚΑΠ είναι η απλούστευση. Τι θα συμβεί όμω με το greening. Αν δεν έχουμε ορατά και αισθητά αποτελέσματα, θα είναι μια απλώ επιπλέον επιβάρηση. Γιατί ε, παρόμοιου στόχου έχει και η πολλαπλή συμμόρφωση. Οπότε το greening δεν είναι καν καλό για τους αγρότες, γιατί τους επιβάλλει επιπλέον υποχρεώσεις για τις ίδιες δραστηριότητε που είχαν και στο παρελθόν. Νομίζω ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις ε, περιστράφηκαν γύρω από τους στόχους ε, του ε, οικολογικού προσανατολισμού. Αλλά δεν μπορώ να σα απαντήσω γιατί αυτό ήταν και το βασικό πόρισμα για διαπίστωση τη δική μα έκθεση. ότι δεν έγινε σαφή προσδιορισμός των στόχων. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ε, το έγγραφο αυτό υποβάλλεται πρώτα στην Επιτροπή Γεωργίας, γιατί η Επιτροπή Γεωργίας διαφορετικά προσεγγίζει αυτό το θέμα και το εξετάζουμε υπό τη σκοπιά περισσότερο και υπό το πρίσμα του γεωργού, αλλά και υπό το πρίσμα του περιβάλλοντος, των σκοπών, των αποτελεσμάτων. Δεν ε, αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα μόνο από τη οικονομική σκοπιά όπως κάνει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, εμείς υθετούμε και άλλες προσεγγίσεις. Οπότε είναι λογικό να διαφέρουμε. Δεν ήμουν χθε στη συζήτηση, προσπαθώ να συμμετέχω στις συνεδριάσεις και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Γεωργίας, γιατί έχω την αίσθηση ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ε, όντως προσπαθεί να εξοικονομήσει τα χρήματα των φορολογουμένων και να πιάνουν τόπο και αυτό είναι θεμητό, αλλά δεν ε, λαμβάνει υπόψη μερικές ιδιαιτερότητες και είναι, φαίνεται πολύ αυστηρή μερικές φορές η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Ε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν ισχύει ότι επειδή έχουμε 27 28 χώρες μέλη έχουμε 28 διαφορετικές γεωργικές πολιτικές. Οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι ενιαίοι. Ο τρόπος εφαρμογής ε, των στόχων είναι ίσως διαφορετικός, γιατί η γεωργία σε κάθε χώρα είναι διαφορετική. Επηρεάζεται από ε, μετερολογικές ε, ε, συνθήκες, από το περιβάλλον, από τις γεωργικές παραδόσεις, από το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, από πολλούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την διακριτική ευχαίρεια των χωρών ή την ελαστικότητα για το τι μέτρα θα επιλέξουν. Γιατί κάθε χώρα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της δικής της γεωργίας. Και γι' αυτό μιλούμε για επικουρικότητα. Αλλά επικουρικότητα δεν σημαίνει επανεθνικοποίηση. Όχι. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της ΚΑΠ, επειδή υπάρχουν και διαφορετικά είδη γεωργίας. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε νέους στόχους, τους ίδιους στόχους. Και ο τρόπος υλοποίησης είναι διαφορετικός. Δεν είναι ότι οι γεωργοί της νότια Ευρώπη δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον ή τη Βόρεια δεν ενδιαφέρονται για το κλίμα. Δεν ισχύει. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν παντού κάποιοι αγρότες που παραβιάζουν τις διατάξεις και δεν σέβονται τις προδιαγραφές. Αλλά αυτό είναι εξαίρεση και ισχύει σε όλους τους κανόνε, σε όλου του κλάδου, συγγνώμη. Ίσως θα μπορούσα να το με η πλάνη της επιτροπης ελεγχου προυπολογισμου γιατι γινονται μερικα λαθη και υπαρχουν μερικες πλαν υπαρχει μερικες φορες μεγάλος ο γεωρικός προϋπολογισμός και δεν εξυπηρετεί και τους στόχους της ΚΑΠ αλλά μερικές φορές έχει λάθος απόψη η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ότι ε, δίνονται χρήματα υπερβολικά για τους νέους γεωργούς και δεν έχουμε αρκετούς νέους γεωργούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν αρκετά τα χρήματα για να μην έχουμε μεγαλύτερο αριθμό νέων γεωργών και δεν μπορούμε να τους προσελκύσουμε. Οπότε έχω και εγώ επιχειρήματα για να καταρρύψω τις, τα επιχειρήματα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Δυστυχώς εκτός μικροφώνου τα σχόλια της κυρίας θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Η κυρία Νόιχλ. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε και η κυρία Κάντεμπαχ. Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Την εκτιμώ και τη σέβομαι. Αλλά το έχετε παρουσιάσει πολλές φορές ως απόψη της ομάδος, της Επιτροπής. Εσείς εκφράζετε την δική σας προσωπική άποψη. Έχετε κάθε δικαίωμα, είσαστε βουλευτής, αλλά δεν είναι αυτή η δική μας άποψη και τοποθέτηση. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να τοποθετούμαστε διαφορετικά. Δεν έχετε το δικαίωμα να συνοψίζετε έτσι την άποψη της Επιτροπής ε, Γεωργίας, γιατί εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις. Εγώ είπα ότι τη δική μου άποψη εκφράζω και τις προσωπικές μου παρατηρήσεις παρουσίασα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει διαφορά απόψεων, καταθέτουμε τροπολογίες και ψηφίζουμε και βγαίνει η στάση της πλειοψηφίας. Αλλά ε, ε, η υπερβολική οικολογικοποίηση δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν ε, εξυπηρετεί την πολωνική γεωργία. Ο κύριος Φλάναγκαν. Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση όταν λέτε ε, εμείς. εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι είναι λαθασμένη η δήλωσή σας. Λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τους αγρότες. Σύμφωνο 100% με τη δήλωση αυτή. Και θα ήθελα πιο πολλούς πόρους και μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να τα πανάτε για τη Γεωργία. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον υπερσμό στόχο. Ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα τροφίμων για τους πολίτες της Ευρώπης. Αν θέλουμε όμως να προστατεύσουμε τους ε, αγρότες, θα πρέπει να ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι εκτός ε, της Επιτροπής μας και όχι να στοχεύουμε τον αγγελιοφόρο και να ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας. Ε. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε με τα σχόλια αυτά, αλλά αν τα αμελήσουμε, μόλις βγούμε από την Επιτροπή αυτή, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα και για τους αγρότες. Αν ακούσουμε, λοιπόν, εγώ ε, θέλω να εκπροσωπήσω τους αγρότες. Ε, για κάθε email που παίρνω όμως από γεωργούς ε, για την ευκρίνηση της ΚΑΠ, παίρνω δύο email για άτομα, από άτομα που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί καν ΚΑΠ και γιατί παίρνουν οι αγρότες τελικά παίρνουν τα χρήματα αυτά. Τους εξηγώ, τους εξηγώ ότι αυτά τα χρήματα τελικά σε εσά επανέρχονται στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες. Αλλά θα πρέπει να ακούμε και να εισακούμε τι λέει ο κόσμος. Λέμε ότι θα πρέπει να ορίζουμε στόχους. Βέβαια, να του ορίσουμε τους στόχους, γιατί το ελεκτικό συνέδριο δεν φαίνεται να ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι μα. Θα πρέπει να του πούμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Γι' αυτό και προσπαθώ να πηγαίνω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού όταν συζητώνται γεωργικά θέματα και στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για να τους εξηγώ τι ιδιαιτερότητε τη γεωργία. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Ο κύριο Χόισλινγκ. Για μένα το θέμα είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον με το ελεκτικό συνέδριο, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα. Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι κανονικά άμα έπρεπε να είναι εδώ και δεν έρχονται. Ο Άλμπερτ βρίζει ωραία ωραία το ελεκτικό συνέδριο και μετά φεύγει. Ε, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να απολογηθούμε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τις εκθέσεις σας μόνο εφόσον μας ταιριάζουν και μας αρέσουν και άμα δεν μας αρέσουν να μην τις αναγνωρίζουμε. Συνάδελφοι και πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει και στους συντονιστέ και έχουμε συναντήσει με το ελεκτικό συνέδριο. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να γίνεται διάλογο, αλλά πολύ απλά δεν μπορεί να επαναληφθεί το σημερινό. Είπατε και δίκαια ή το είπατε ότι αυτή την εντολή μας δώσατε και δεν μπορούμε παρά να παρουσιάσουμε αυτά που βρήκαμε. Ε, προφανώς, δίκιο έχετε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε τα ευρήματα και τα πορίσματα εν ώψη της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ προφανώς. Δεν μπορούμε απλά να μην τα λάβουμε υπόψη. Εμείς λοιπόν ε, ε, νομίζω ότι ξεχάσαμε τα πορίσματα της έρευνας αυτής και τα σε ευχαριστώ. Συμφωνώ. Ανέκαθεν ε, επενούσα και έλεγα πόσο εκτιμούμε τις απόψεις του ελεκτικού συνεδρίου και πόσο εκτιμούμε την προσπάθεια του ελεκτικού συνεδρίου. Και μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές απόψεων, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προσβάλλουμε ή να είμαστε τόσο απότομοι απέναντι στο ελεκτικό συνέδριο. Κύριε Μπογκόβιτς. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι δεν συμπίπτουν απόλυτα οι απόψεις μας. Και εγώ δεν συμφωνώ με την παρατήρηση ότι τίποτα δεν αλλάζει στη Γεωργία γιατί εγώ γεννήθηκα σε μια φάρμα και ασχολούμαι με τη γεωργία από το 1984 και ξέρω πόσα άλλαξαν στην Σλοβενική Γεωργία μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ, στην Επιτροπή Γεωργίας, δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι οι γεωργικές πρακτικές είναι πολύ πιο ευνοϊκές και πολύ πιο φιλοπεριβαλλοντικές από ό,τι στο παρελθόν και φυσικά είναι κοινό μας καθήκον να βελτιώσουμε περαιτέρω και στο μέλλον αυτές τις γεωργικές πρακτικές για να γίνουν ακόμη πιο φιλοπεριβαλλοντικές. Αν όμως ε, μιλάμε τόσο αρνητικά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και ότι άδικα παίρνουν τι ενισχύσει οι γεωργοί, πώς είναι δυνατόν να διαφυλάξουμε τον γεωργικό προϋπολογισμό αν μιλούμε έτσι περιφρονητικά για τη Γεωργία. Θεωρώ ότι έχουν, έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος και θα πρέπει να είμαστε ευρηματικοί και να βρούμε ε, δημιουργικές λύσεις, ώστε και να κρατήσουμε τα κονδύλια της γεωργίας και να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ασχοληθούν ε, με τη γεωργική δραστηριότητα ή να παραμείνουν στη γεωργία αν έχουν ξεκινήσει. Και φυσικά δεν μπορώ να συμφωνήσω στα πάντα, αλλά και στο θέμα του οικολογικού προσανατολισμού του Greening